Ε, θα κατατεθούν ε, στο Κοινοβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν σήμερα ε, θα τα διαβιβάσω στους αρμόδιους. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση και εύχομαι σε όλους σας καλή επιστροφή στα σπίτια σας και καλό Σαββατοκύριακο.